Ε, προσωπικών δικαιωμάτων, την ελευθερία της, ε, της, της, της των θρησκευτικών στο Πακιστάν και παντού. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ. Έχει λήξει η συζήτηση για το θέμα του Πακιστάν. Έχω 7 προτάσεις ψηφισμάτων και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία όταν ολοκληρώσουμε τις άλλες δύο συζητήσεις. Η επόμενη είναι θέμα για την Βραζιλία έκδοση του Τσέζαρη Μπατίστη. Εδώ υπάρχουν έξι συντάκτες του, της προτάσεως ψηφίσματος. Πρώτη θα λάβει τον λόγο η κυρία Μπιζόνα. Για το διεθνές δίκαιο θεωρείται πολιτικός πρόσφυγας αυτός ο οποίος διώκεται λόγω φιλής, κοινωνικής, ε, πολιτικής ε, ή πολιτικού ανήκειν. Ο Τσέζαρε Μπατίστη δεν είναι πολιτικός πρόσφυγας. Παρά την κάλυψη που του έχει δοθεί από τη Γαλλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένας εντολοδόχος δολοφονιών. Τέσσερις δολοφονίες έχει διατάξει. Είναι καταδικασμένος σε ισόβια δεσμά. Η Βραζιλία αντιστέκεται στην έκδοση ενός δολοφόνου. Οι Ιταλικές αρχές και οι οικογένειες των θυμάτων θέλουν να παραδοθεί στην δικαιοσύνη αυτός ο φυγάς. Ο κύριος Λούλα όμως αρνείται. Η Ιταλική κυβέρνηση δεν θα πρέπει να είναι μόνη της για να αντιμετωπίσει το αίτημα το αίτημά της. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πιέσει ακόμη και σταματώντας, παραλύοντας τις ε, συμφωνίες με την Βραζίλια. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, το κράτος του δικαίου, είναι βασικές έννοιες της δημοκρατίας στις δημοκρατικές τουλάχιστον χώρες. Κάθε εξωπρεπές, ε, κάθε πολίτης ε, έχει το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη. Τα ανεξάρτητα δικαστήρια λοιπόν πρέπει να γίνονται σεβαστά. Σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο δικαστήριο στη Βραζιλία έχει λάβει μια απόφαση που επιτρέπει την έκδοση του Τσέζαρε Μπατίστη στην Ιταλία. Η Ιταλία αποφάσισε να ζητήσει την έκδοσή του βάσει των κανόνων και των ρυθμίσεων που ήδη ισχύουν. Και το Διεθνές Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έλαβε υπόψη την προσφυγή της χώρας αυτής. Το ζήτημα κανονικά έχει επιληθεί. Βρισκόμαστε στο τέλος της υπόθεσης αυτής. Αυτή τη στιγμή πρέπει η Βραζιλία να δράσει κατά τρόπον ώστε η δικαιοσύνη να ε, μπορέσει να γίνει σεβαστή. Δηλαδή να γίνει η έκδοση. Ελπίζω ότι η υπηρεσία εξωτερικής δράσης θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το κάτω δικαίου γίνεται σεβαστό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρωμέβα ε, Ιρουέδα για δύο λεπτά. Εγώ να μην ε, σας ε, το αποκρύψω ότι αισθάνομαι αμήχανος με το θέμα και με την κατάσταση διότι έχουμε ένα θέμα σημαντικό το οποίο αφορά στην Ιταλία και στην Βραζιλία και υπάρχουν πολλοί χώροι για τους, μέσα στους οποίους μπορεί να συζητηθεί το θέμα αν εδώ είναι ο κατάλληλος χώρος για να γίνει η συζήτηση και κατά την ώρα της συζήτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εγώ εκφράζω την απόλυτη αλληλεγγύη μου στα θύματα της τρομοκρατίας όπου και αν βρίσκονται και με τα θύματα στη συγκεκριμένη υπόθεση. Εγώ απλώς εδώ θέλω να τονίσω πως θέματα τόσο σοβαρά έρχονται την πέμπτη το απόγευμα. Έχουμε μια κατάσταση σουπιούντισε, ήδη δεδικασμένη, και μια διαδικασία έκδοσης η οποία έχει ξεκινήσει. Εμείς θα απόσχουμε, όχι γιατί το θέμα δεν πρέπει να το σκεφτούμε, αλλά απλώς θεωρούμε ότι δεν είναι ούτε η ώρα ούτε ο τόπος για να συζητηθεί το θέμα. Κυρία Αντζελίλη. Με αυτό το ψήφισμα απευθύνουμε έκκληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα τα οποία κατά την άσκηση των διπλωματικών τους δραστηριοτήτων να παίξουν ένα ρόλο για το σεβασμό της δικαιοσύνης και της νομιμότητας. Το Κοινοβούλιο σήμερα ζητά η Χάρτα των Δικαιωμάτων να μην είναι απλώς ένα χαρτί να μην είναι μόνο καταναλωτές μιας κοινή αγοράς οι πολίτες αλλά δικαιούχοι θεμελιωδών και απαραβιάστων δικαιωμάτων. Με αυτό το πνεύμα εμπιστοσύνης ε, ήταν εδώ παρόντες ε, τέσσερις ε, από τις τέσσερις οικογένειες των θυμάτων του Μπατίστη θύματα τα οποία δολοφονήθηκαν ψυχρά μπροστά στις οικογένειές τους και στα παιδιά τους. Εμείς ε, τρέφουμε εμπιστοσύνη στο δίκαιο και σας παρακαλώ να κρατήσουμε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων. Ο κύριος Σασόλη. Εμείς είμαστε σήμερα εδώ στην Ολομέλεια για να θυμίσουμε πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα, ε, δημοκρατικά θεσμικά όργανα θα πρέπει να βρίσκονται κοντά στις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας και να δίνουν και ένα νόημα σε, σε αυτό το αίσθημα δικαιοσύνης που απαιτεί η κοινωνία. Στο ψήφισμα που θα ψηφίσουμε λέμε ότι υπάρχει αμοιβαία αναγνώριση και σεβασμός μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βραζιλίας. Δεν υπάρχει κανένα θέμα που να υποσκάπτει τις χιλικές σχέσεις με τη Βραζιλία. Ο Τσέζαρε Μπατίστη στην Ιταλία καταδικάστηκε για τέσσερις δολοφονίες και ακόμη και παράνομος όντας είχε όλες τις νομικές εγγύησεις κατά τις δίκες του δικάστηκε δίκαια παρουσία του δικηγόρου του και η Ιταλική δικαιοσύνη σεβάστηκε όλες τις, όλα τα δικαστικά επίπεδα και έχει καταδικαστεί σε διπλά ισόβια δεσμά. Και στη Γαλλία η Γαλλία όπου κατέφυγε ο, διέφυγε ο Μπατίστη είχε δεχθεί το 2004 να τον, απελάσει, να τον εκδώσει στην Ιταλία έχοντας αναγνωρίσει και, τη, και τα εγκλήματά του και τις δύο καταδίκες του είναι ένας καταδικασμένος πρέπει να εκδοθεί να δοθεί στη δικαιοσύνη δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η Βραζιλία δεν το αναγνωρίζει αυτό γιατί οι, Βραζιλι... οι αρχές της Βραζιλίας δεν το έχουν αναγνωρίσει το καθεστώς του πολιτικού πρόσφυγα Γι' αυτό μας φάνηκε, φάνηκε ακατανόητη η απόφαση του Ανωτάτου Βραζιλιανικού Δικαστηρίου στα, στις οικογένειες των θυμάτων. Είμαστε οι εκπρόσωποι της Ευρώπης των δικαιωμάτων όλων και θα πρέπει οι καταδικασμένοι να εκτίουν τις ποινές τους στις φυλακές των χωρών τους. Κύριος Τσαρνιέσκη. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, εγώ ούτε Ιταλιάνος είμαι, Ιταλός είμαι, ούτε Βραζιλιάνος. Εγώ είμαι ένα μέλος, ένας πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα ήθελα να έχουμε μια συμμετρική Ευρώπη όπου τα ίδια δικαιώματα τα παρέχουμε στα θύματα και στους θύτες. Είναι ένα θέμα απαράδεκτο για μένα. Ε, θεωρώ ότι δεν είναι ανθρώπινο κάτι τέτοιο. Όταν ε, επειδή εγώ δεν τρέφω ιδιαίτερα συγκινησιακό, δεν έχω ιδιαίτερη συγκινησιακό φόρτο σε αυτό το θέμα, πρέπει να σας πω ότι πρέπει να βρούμε μία ισορροπία που, ισορροπία που είναι σημαντική για τους πολίτες που μας ψηφίζουν και τους φορολογούμενους. Αυτό το θέμα με τη Βραζιλία είναι πραγματικά αδιανόητο. Δεν μπορεί να το κατανοήσει κανένας Ευρωπαίος πολίτης. εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων ο Μάριο Μάουρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εχθές σε μία συνέντευξη τύπου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οικογένειες των θυμάτων έθεσαν πάλι το φόντο αυτής της δραματικής υπόθεσης όχι βεντέτα, όχι εκδίκηση, αλλά δικαιοσύνη. Και για να αποδοθεί δικαιοσύνη πρέπει να εκδοθεί ο Μπατίστη. Και για να εκδοθεί ο Μπατίστη ε, θα θέλαμε με αυτό το ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να είναι ο να, είναι η αντίχηση αυτής της κραυγής ότι πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη και όχι εκδίκηση. Η Ευρώπη είναι ένα πολιτικό σχέδιο όπου θέσαμε από κοινού αξίες ε, και ιδανικά για να γκρεμίσουμε τον βαρβαρισμό των απολυταρχικών ιδεολογιών, την άβυσο του κακού και της τρομοκρατίας. Για να ολοκληρώσουμε αυτό το σχέδιο ζητάμε δυναμικά σήμερα. Καμία εκδίκηση, αλλά να αποδοθεί δικαιοσύνη. Ευχαριστώ για τους σοσιαλιστές ο κύριος Σούστα. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι βουλευτές, κύριε Επίτροπε, τυχαίνει συχνά διανοούμενοι οι θεσμοί άλλων χωρών να αρνούνται να καταλάβουν το φαινόμενο της Ιταλικής τρομοκρατίας αμφισβητώντας ε, την αξιοπιστία του δικαστικού μας συστήματος. Αυτή είναι και η νομική προϋπόθεση για την άρνηση της έκδοσης του Μπατίστη και το απορρίπτουμε. Ο Μπατίστη με αμφισβητούμενα προηγούμενα είναι καρπός μιας εποχής όπου μοναχικοί και απελπισμένοι νέοι τόριξαν στον ένοπλο αγώνα και κατέληξαν στο γκρέμισμα της ουτοπίας των πιστεύων τους. Και σε άλλες χώρες συνέβησαν τα ίδια. Καμιά όμως δεν έδωσε τις ευκαιρίες που έδωσε η Ιταλία, η οποία μέσα από την καταπολέμηση της τρομοκρατίας θεμελίωσε και το αίσθημα της εθνικής της ενότητας. Θέλουμε εμείς ο Μπατίστη να αποδοθεί στην Ιταλική δικαιοσύνη. Διαπιστώσατε ότι υπάρχουν χιλιάδες πρώην τρομοκράτες οι οποίοι έχουν επανεισέλθει στην κοινότητα στην ε, κοινότητα. Ο Μπεκαρία μιλούσε για την, για τον, την τιμή της ποινή και την αναλογικότητα. Εκ της κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Εδώ ασχολούμαστε με ένα θέμα που δεν είναι πραγματικά κατεπήγον. Όμως Νομίζω ότι κατά κατεπήγοντα θα είχαμε πολύ σοβαρά θέματα να συζητήσουμε, όπω ο φυλακισμό και τα βασανιστήρια κατά των συνδικαλιστών στην ε, Κολομβία, το τι συμβαίνει στι Ονδούρες ή στα κατεχόμενα τη Παλαιστίνη από το Ισραήλ. Ε, εάν θέλουμε να μιλήσουμε για τη Βραζιλία, ε, Α σκεφτούμε αν πρόκειται για αληθινά κατεπήγον και το τι συμβαίνει με τους πληθυσμούς που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Και ε, που έπληξαν το κράτος, το κρατήδιο του Ρίο Ντετζανέιρο ε, της Τερεζόπολης ε, και που προκάλεσαν εκατοντάδες θανάτους άφησαν άστεγους πολλούς ανθρώπους και πολλούς τραυματίες. Αυτή είναι μια πραγματική τραγωδία για την οποία δεν αποφάνθηκε η το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε διέθεσε την απαραίτητη βοήθεια για να στηρίξει αυτή τη χώρα. Χαιρετίζουμε λοιπόν την ε, δράση της νέας Πρόεδρου της Βραζιλίας, της Ντίλμα Ρουσέ, που ελπίζουμε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί και εκφράζουμε την αλληλεγγύη, της, την αλληλεγγύη μας για να αντιμετωπίσει ακριβώς την δύσκολη αυτή κατάσταση με τα θύματα των πλημμυρών. Ε, ελπίζουμε ότι το ε, βραζιλιανικό κράτος θα καταφέρει να καλύψει τα θύματα της τραγωδίας αυτή και των οικογενειών τους η ε, ε, περίπτωση αυτή τώρα νομίζω ότι δείχνει την ανάγκη να σεβαστούμε τα, ε, τις αποφάσεις των επισήμων δικαστικών οργάνων της Βραζιλίας που είναι δημοκρατικά εκλεγμένα και που έχουν τοποθετηθεί σε σχέση με την περίπτωση του κυρίου Μπατίστη. Θα έλεγα λοιπόν να μην λάβουμε εδώ μία απόφαση που μετά θα μας δυσαρεστήσει. Σας ευχαριστούμε. Ο ο κύριο Περόνη σήκωσε την κενή του κάρτα. Να ρωτήσω τη συνάδελφο που είπε ότι υπάρχουν τόσα πολλά κατεπήγοντα. Το εξή. Διαφορετικά από άλλες καταστάσεις που σίγουρα είναι κατεπήγον, κατεπήγουσες, αυτό είναι ένα κατεπήγον το οποίο εμπλέκει όχι μία χώρα εκ των έξω αλλά και μία χώρα εκ των έσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναφερόμαστε εδώ σε πολίτες οι οποίοι δολοφονήθηκαν ή έμειναν ανάπηροι και είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Κυρία Φιγκερέη, που θέλετε να απαντήσετε. Μα το είπα ήδη και θα το επαναλάβω. Εδώ δεν έχουμε πραγματικά ένα κατεπήγον ζήτημα. Ξέρουμε ότι τα επίσημα, οι επίσημοι φορείς της Βραζιλίας εξετάζουν την περίπτωση αυτή. Και ο πολίτης αυτός κρατείται στην Βραζιλία. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν μπορεί να ασκήσει πιέσει ε, κατά των επισήμων φορέων και οργάνων τη Βραζιλία. Πρέπει να σεβαστούμε τι αποφάσει του ή τις αποφάσεις που θα λάβουν ε, στο μέλλον για τα κατεπήγοντα έχουμε να συζητήσουμε πολλά άλλα θέματα που πάλι μπορεί να αφορούν τη Βραζιλία. Την αλληλεγγύη που θα πρέπει να εκφράσουμε στα θύματα, τα θύματα των καταιγίδων, των πλημμυρών με τους 700 νεκρούς που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία. We have, we have blue card, Έχουμε και άλλη γαλαζιά κάρτα από την κυρία Αντζελίλη. Απλή ερώτηση στην κυρία Φιγκερέιδο ε, δεν νομίζετε ότι 30 χρόνια, γιατί 30 χρόνια πέρασαν από τη δολοφονία αυτών των ανθρώπων, αν αυτά τα 30 χρόνια δεν αρκούν, ούτως ώστε πλέον κατεπηγόντως να ζητήσουμε την απόδοση της δικαιοσύνης. Η κυρία Φιγκερέιδο. Ήδη το είπαμε. Να το επαναλάβω κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά το θέμα είναι ο τρόπος, το πλαίσιο εντός του οποίου συζητάμε το θέμα αυτό. Το συζητάμε τη στιγμή του προγράμματος ότι πρέπει να συζητήσουμε τα κατεπήγοντα ζητήματα. Μόλις το είπατε κι εσείς, συνάδελφε. Είναι σαφές το θέμα αυτό μπορούσαμε να το είχαμε συζητήσει τόσες άλλες φορές. Και έτσι θα έπρεπε να γίνει. Αυτή τη στιγμή, τη στιγμή των κατεπηγόντων, δεν είναι κατάλληλη η στιγμή. Να εκφράσουμε την ελληνική μα για τα 700 θύματα τη τραγωδία τη Βραζιλία τι τελευταίε ημέρε, με τι πλημμύρε και τι καταιγίδε. Ευχαριστούμε. Καταλάβαμε τι λέτε. Να ακούσουμε τώρα τον επόμενο μιλητή μα, τον κύριο Προβέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο Τσέζαρε Μπατίστη δεν είναι ένα ρομαντικό ήρωα, αλλά ένα όπως κάτι τον περιέγραψαν, αλλά ένας άγριος ε, δολοφόνος, ο οποίος έχει κάνει κλοπές και έχει καταδικαστεί γιατί σκότωσε ε, εν ψυχρό τέσσερα άτομα. Εποφελήθηκε από το δόγμα Μιτεράν για το πολιτικό άσυλο και προστατεύθηκε και κάποιες φορές αγιοποιήθηκε από κάποιους διανοούμενους της γαλλικής αριστεράς. Διέφυγε στη Βραζιλία για να αποφύγει την ε, αναπομπή του στη χώρα, και την, στη χώρα του και την ε, φυλάκισή του και διασώθηκε από τον πρόεδρο Λούλα βάσει μια ασφαλμένη απόφαση. Ίσως για πολιτικού λόγου και χωρί να ληφθεί υπόψη ο πόνο των θυμάτων των οικογενειών και των οικογενειών. Η έκκληση του Κοινοβουλίου μα προ τι Βραζιλιανικέ Αρχέ και την Επιτροπή δεν ζητά μόνο να γίνουν σεβαστοί οι νομικοί κανόνε και οι διμερεί ε, συμφωνίε, αλλά να μην χρησιμοποιείται καμία ιδεολογική αρχή ω πρόσχημα για να προστατεύεται ένα δολοφόνο και να μην εξασφαλίζει την ατιμορρυσία του κανένα κράτο. Να μην ξεχνάμε ότι εδώ θα πρέπει να, από ηθικής άποψης να εξασφαλίσουμε ηθική ικανοποίηση στα θύματα και βάσει του κοινωνικού συμβολέου που ουσιαστικά βρίσκεται στα θεμέλια οποιασδήποτε κοινωνίας πολιτών που θέλει έτσι να ονομάζεται. Ευχαριστούμε κύριο Γιακολίνο. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τόσα χρόνια μετά το αίμα των ε, θυμάτων ε, των βάρβαρων δολοφολιών του Τσέζαρε Μπατίτη και της συμμορίας του ε, δεν το έχουμε ξεχάσει. Οι οικογένειες που ακούσαμε χθε να εκφράζονται στην συνέντευξη τύπου στο Στρασβούργο είναι μια πραγματική απόδειξη. Το είπε ο συνάδελφος Μαστέλα που ήταν τότε υπουργό δικαιοσύνη στην Ιταλία είχε καταβάλει σκληρές προσπάθειες με θεσμικές ε, δράσεις προκειμένου να αποδοθεί δικαιοσύνη στην υπόθεση Μπατίστη. Σήμερα ε, μεταξύ των ε, θυμάτων και των οικογενειών τους και σε όλη την κοινωνία της Ιταλίας θα πρέπει να αποδείξει το Ευρωκοινοβούλιο ότι μπορεί να είναι αλληλέγγυο με την πρόταση αυτή ψηφίσματος να ζητήσει με ένταση από μια άλλη χώρα φίλη της Ευρώπης, φίλη της Ιταλίας αμέσως να εκδώσει τον Τσέζαρε Μπατίστη. Είναι εγκληματίας, είναι τρομοκράτης και έχει καταδικαστεί με ποινές ε, στο παρελθόν. Για να ολοκληρώσω η θλιβερή αυτή υπόθεση εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν έχει κάποια λύση. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε τώρα. Ευχαριστούμε. Catch the eye τώρα. Συνάδελφοι, έχω περίπου 20 ονόματα στον κατάλογο μου. Γαλάζια κάρτα ή κάτι άλλο. Έχετε γαλάζια κάρτα για τον προηγούμενο μιλητή. Ή... Ε, είναι, σηκώνετε γαλάζια κάρτα γιατί θέλετε να ρωτήσετε τον προλαλήσαντα. Έχει καλώς. Δεν είναι λοιπόν αυτή η περίπτωση. Καλά. Έχω το πρόβλημα ότι έχω 20 εγγεγραμμένους ομιλητές όμως αυτή τη φορά θα δώσω το λόγο μόνο στα πρόσωπα εκείνα τα οποία δεν μπόρεσαν να μιλήσουν πριν στο, για το Πακιστάν δηλαδή. Ελπίζω ότι το δέχεστε αυτό. Πρώτα, Φιντάντσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από μόνος του ήταν ένας μικροεγκληματίας, ε, αλλά πολύ ξύπνιος. Και αποφάσισε να γίνει και πολιτικός. τα θύματα τα οποία επλήγησαν σωματικά και ψυχικά από την ομάδα του δεν ζήτησαν ποτέ εκδίκηση. Ζήτησαν δικαιοσύνη. Όχι γιατί είχε την απόφαση, την καταδίκη για τα ισόβια. Απλώς Απλώς θέλουν δικαιοσύνη. Αυτό λέει για, για τον Τσέζαρε Μπατίστη, ο Καβαλίνα που ήταν αυτός που τον οστρατολόγησε στην πολιτική έχει καταδικαστεί ο Μπατίστη για τέσσερις δολοφονίες. Πρώτα διέφυγε στο Μεξικό, μετά στη Γαλλία και τώρα στη Βραζιλία και τον περνάνε για ρομαντικό επαναστάτη και όχι για έναν άσπλαχνο εκτελεστή. Η κατάσταση λοιπόν στο, η υπόθεση του Μπατίστη στην Ιταλία δεν είναι αυτό που κάτι διανοούμενοι σαλονιών θέλουν να μας κάνουν να πιστεύουν ότι είναι ένα θέμα εκδίκησης. Όχι, είναι θέμα σεβασμού των διεθνών συνθήκων και των δικαστικών άρχων. Ο κύριος Στάνοκ. Εγώ δεν συμφωνώ ότι πρέπει να δώσετε το χρόνο ομιλία στο ΚΑΤΣΤΙΑΙ σε σχέση με το ποιο παρενέβη για το Πακιστάν. Είναι τελείω διαφορετικό το ζήτημα αυτό. Εδώ κάποιοι χάνουν το χρόνο του στα τηλέφωνα, ίσω γι' αυτό να μην ήταν προηγουμένω στην αίθουσα. Λοιπόν, είναι θέμα αντιπροσωπιών και πολιτικών ομάδων και ίσω κάποιοι να ωφεληθούν. Θα συμφωνήσω μαζί σα ότι πρόκειται για τελείω διαφορετική συζήτηση, αλλά έχουμε δώσει δύο λεπτά. Άρα έχω δυνατότητα να δώσω το λόγο σε δύο πρόσωπα. Τι θα κάνατε αν ήσασταν στη θέση μου. Εγώ θέλω πολύ ευχαρίστω να δώσω ισότιμα το λόγο σε όλους όσοι δεν μίλησαν πριν σε όσους μίλησαν πριν σε κάθε εκπρόσωπο πολιτική ομάδα. και γνωρίζω βεβαίω ότι μίλησαν κατ' εξοχήν οι Ιταλοί συνάδελφοί μας τώρα ακολουθεί η κυρία Κόρφολα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε Αντιλαμβάνομαι την απογοήτευση των συναδέλφων όταν μιλούν για τον κατεπήγοντα χαρακτήρα του κειμένου. Όταν ο πρόεδρος Λούλα αποφάσισε να μην εκδώσει τον Μπατίστη, ανακάλεσε τον πρέσβη του ο πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη για να ζητήσει ξανά με περισσότερη έμφαση την έκδοση. Γίνεται αγώνας. Ένας αγώνας που έχει κρατήσει 30 χρόνια μεταξύ των διαφορών οργάνων δικαιοσύνης. Κανονικά θα ήταν στην φυλακή αυτός για εσόβια. Εμείς, εάν θεωρηθεί κάποιος κατάδικος ως πολιτικός κρατούμενος, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ορθό αυτό. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο, please. Consider că respectarea independenței justiției e norma fundamentală împărtășită de Uniunea η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί θεμελιώδη αρχή, την οποία σέβονται και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βραζιλία. Και αυτή πρέπει να κυριαρχήσει. Είμαι βεβαία ότι οι θαυμάσιες σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών θα οδηγήσουν και σε καλή συνεργασία των οργάνων δικαιοσύνης ώστε ο Μπατίστη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για τέσσερις φόνους, εν τέλει να εκτίσει την ποινή του. Υπάρχουν και, υπάρχει μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας και διμερή συμφωνία εκδόσεως. Ωστόσο, έχει και υψηλή πολιτική σημασία ε, η περίπτωση αυτή και πρέπει να συζητηθεί με τη νέα Βραζιλιάνα Πρόεδρο. Η κυρία Βερζιάν. Ε, πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εμένα με εκπλήσει το πόσο πολλοί βουλευτέ βρίσκονται παράντως σε αυτό το ημικύκλιο πέμπτη απόγευμα. Εγώ είμαι εδώ κάθε πέμπτη απόγευμα και βρίσκω ότι αυτή η παρουσία δείχνει ένα τεράστιο ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι ένα έκτακτο γεγονό αυτό. Θα ήθελα όμω να συγχαρώ όσου κάνουν τέτοια βήματα, ιδίω του Ιταλού βουλευτέ που βρίσκονται σήμερα στην αίθουσα τη Ολομέλεια. Συνήθω δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πολύ συχνά φαίνεται να έχουν ελλημένες υποχρεώσεις Θέλετε να εκφραστείτε, αγαπητέ συνάδελφοι, κάνετε στο μικρόφωνο και θα σας απαντήσω. Ε, μπορεί να είναι και προσωπική η συζήτησή μα. Είστε Ιταλό είμαι Γαλλίδα. Ε, εγώ σέβομαι, μάλλον παρατηρώ το τι συμβαίνει με του ε, Ιταλού συναδέλφου. Εδώ είναι πλειοψηφία. Αυτό συνήθω είναι ασυνήθιστο για τι Πέμπτε το απόγευμα. Εγώ είμαι εδώ κάθε Πέμπτη απόγευμα, αγαπητέ μου κύριε, εντάξει. Κάθε Πέμπτη απόγευμα είμαι στην Ολομέλεια. Αφήστε μου να μιλήσω. Πρόεδρος, παρακαλώ, συνάδελφοι, ησυχία. Εγώ δεν διέκοψα του συναδέλφου, δεν δέχομαι να με διακόπτουν. Μπορώ να συνεχίσω, Πρόεδρε. Ε, βλέπω λοιπόν ότι ενώ γενικώ οι Ιταλοί συνάδελφοι είναι οι πρώτοι που, διερωτών, που ζητούν μάλλον να μην γίνεται ανάμειξη στι εσωτερικέ υποθέσει τη Ιταλία, ε, δεν συμμετέχουν σε τέτοιε συζητήσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ το θέμα δεν είναι αν είναι ένοχο ή όχι ο Τσέζαρη Μπατίστη. Γνωρίζω και απευθύνομαι και πάλι σε εσά. Γνωρίζω ότι τα πέτρινα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα για την Ιταλία. Τα χρόνια τα μολύβδινα. Ε, όμως ε, ήταν πολλά τα θύματα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλοι οι ένοχοι που έχουν διαπράξει απόπειρε δεν έχουν ε, προσαχθεί στη δικαιοσύνη στην Ιταλία. Όσοι έκαναν δολοφονικέ απόπειρε δεν έχουν δικαστεί στην Ιταλία. Παρακαλούμε, έχετε μόνο ένα λεπτό. Μα αφήστε με να μιλήσω, παρακαλώ. Με διακόπτετε συνέχεια. Είστε στο εθνικό σα κοινοβούλιο. Εδώ είναι Ευρωκοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω, θα τοποθετηθώ ή όχι. Έχετε 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσετε την παρέμβασή σα, διότι έχουμε ξεπεράσει τον χρόνο. Με όλε τι διακοπέ. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ τον χρόνο. Νομίζω λοιπόν ότι πέμπτη απόγευμα ε, δεν είναι η στιγμή να συζητήσουμε τι σχέσει Ιταλία και Βραζιλία, αλλά θέλουμε να επιβάλλουμε τον σεβασμό για την δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ. Όμω, α αφήσουμε τον, το δικαστήριο τη Βραζιλία να έχει το χρόνο στη διαθεσία του για να ε, εκδώσει την απόφασή του. Ε, η δικαιοσύνη τη Βραζιλία μόλι ανέλαβε να εξετάζει το θέμα. Δεν έχει τοποθετηθεί. Με συγχωρείτε, πρέπει να σα διακόψω. Πρέπει να σα διακόψω. Έχουμε ένα λεπτό για την διαδικασία αυτή. Μα κοιτάξτε, εγώ ήθελα να μιλήσω για ένα λεπτό, αλλά όχι, όχι, έχετε ξεπεράσει όλου του άλλου συναδέλφου με τρία λεπτά. Εγαλάζια κάρτα από την κυρία Αντζελίλη. μπορώ να μιλήσω χωρίς να με διακόπτουν. Δεν τελείωσα καμία φράση μου. Ένα λεπτό οι παρεμβάσει. Με όλε τι διακοπέ σα έδωσα παραπάνω χρόνο. Κυρία Αντζελίλη, γαλάζια κάρτα. Θα απαντήσετε. Κυρία Βερζιά, θα απαντήσετε. Yes. Okay. Κύριε Πρόεδρε, σέβομαι του συναδέλφου και βεβαίω θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτηση. Αλλά θα ήθελα και οι ίδιοι να δείξουν ανοχή όταν εγώ παίρνω το λόγο. Αν εσεί, κυρία Βερζά σέβεστε τους συναδέλφους δεν θα έπρεπε να επιτρέπετε στον εαυτό σας να λέτε ότι οι Ιταλοί συνάδελφοι δεν ενδιαφέρονται ποτέ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ είμαι μέλος εδώ 16 χρόνια. Ελέγξτε λοιπόν την κοινοβουλευτική μου δραστηριότητα και σίγουρα δεν αξίζω μαθήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων από εσά. Madame Κοιτάξτε κύριε Άντζελη, αυτό που κάνετε ήταν δήλωση. Όταν σηκώνετε τη γαλάζια σας κάρτα σημαίνει ότι θέλετε να κάνετε ερώτηση. Στο όνομα των συναδέλφων θέλαμε να τη ρωτήσουμε αν δεν τρέπετε ή όχι θέλετε να σηκωθείτε αν δεν τρέπεται ή όχι, για αυτούς τους τέσσερις. Αυτοί οι τέσσερις ήταν ο ένας ήταν δικαστικός κλητήρας, ο άλλος ήταν χασάπης, ο άλλος ήταν έμπορος και ο άλλος ήταν χωροφύλακας. Εχθέ τα παιδιά αυτών των τεσσάρων που, ήταν, που είχαν 10, 15 χρονών τότε μας λένε ότι κάθε άγια μέρα της ζωή τους θυμούνται το γονιό τους μέσα σε ένα ποτάμι αίματο. Εσεί θεωρείτε ότι από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε μια πολεμική. Η κυρία Βερζά. Κύριε Πρόεδρε, θεωρώ ότι αυτό το θέμα είναι καθαρά προσωπικό, όχι δεν ντρέπομαι διότι σας είπα ότι θεωρώ τα, χρόνια, τα μολύβδινα χρόνια, δύσκολα χρόνια για την Ιταλία. Σας το είπα. Ξέρω πολύ καλά πόσα θύματα υπήρξαν στην Ιταλία. Ενδιαφέρθηκα προσωπικά για αυτήν την περίοδο. Όχι, δεν τρέπομαι. Δεν αμφισβητώ τα θύματα. Αμφισβητώ την χρήση εκ μέρους των Ιταλών βουλευτών της Πέμπτης της Ολομελίας του απογεύματος που ασχολείται με ανθρώπινα δικαιώματα για να θέσει ένα διμερές θέμα μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παρέμβει στις Ιταλο-Βραζιλιανικές σχέσεις και αυτό μέσα στο timing των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και δεν θέλω να σας δώσω μαθήματα σχετικά. Άλλες δύο μπλε κάρτες. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο μιλητή. Διαδικαστικό, κύριε Μάουρο. Ναι. Λοιπόν, αφορά στο άρθρο εκείνο του κανονισμού που αφορά στην ημερήσια διάταξη. Πρέπει να σας θυμίσω ότι αυτό το σημείο μπήκε στην ημερήσια διάταξη από τη διάσκεψη των Προέδρων και επικυρώθηκε από την Ολομέλεια της Δευτέρας. Δεν είναι κάτι, ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη που μπήκε μετά από κέφι των Ιταλών βουλευτών. Όχι, είναι ένα θέμα το οποίο μπήκε μετά από νόμιμη απόφαση του Κοινοβουλίου. Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, ο κύριος Ρώση, τελευταίος αγορητής. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι εγκύτρια της συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας και Βραζιλίας και να, να γίνουν σεβαστές οι αρχές σχετικά με την έκδοση. Η Ιταλία έχει καταδικάσει σε 7 δίκες ερήμην ε, για τον Μπατίστη. Δύο ε, διπλά ισόβια για τέσσερις δολοφονίες. Ο πρόεδρος της Βραζιλίας αρνήθηκε να παραδώσει τον εγκληματία στην Ιταλία και όχι μόνο. Ιδιαίτερα υποτιμητικά αριστεροί βραζιλιανοί βουλευτές πήγανε στη φυλακή να επισκεφθούν τον Πατίστη και βγήκαν και φωτογραφία γιορτάζοντας την απόφαση. Δεν μπορεί λοιπόν η Ιταλία να μην παρέμβει και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις, μέσα από τις εμπορικές της συμφωνίες να μην παρέμβει για να, γίνει, να αποδοθεί δικαιοσύνη στα θύματα. Εχθέ, οι οικογένειε των θυμάτων ήρθαν στο Στρασβούργο και εχθέ όλοι όσοι ήταν παρόντε και άσχετα από το πολιτικό του ανήκει συμφωνήσανε γύρω από το θέμα. Ο επίτροπο. Uh, Ο Επίτροπος Φίλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόφαση του απερχομένου Βραζιλιάνου Προέδρου να απορρίψει την αίτηση έκδοσης του Τσέζαρε Μπατίστη που έχει καταδικαστεί από τα Ιταλικά δικαστήρια για φόνους και άλλα εγκλήματα. Σημείωσα τις απόψεις που εκφράσατε. Συμμερίζομαι τα αισθήματά σας απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει περιθώριο παρέμβασής της στην υπόθεση αυτή. Δεν έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνία εκδόσεως με την Βραζιλία και αν ακόμα συνέβαινε κάτι τέτοιο δεν θα είχε δικαίωμα να παρέμβει σε μεμονωμένες ατομικές υποθέσεις εκδόσεως. είτε ανάμεσα σε χώρες ε, μέλη, είτε μεταξύ χωρών μελών και τρίτων χωρών. Η σχέση με τη Βραζιλία για την δικαστική αρρωγή σε θέματα ποινική δικαιοσύνης διέπονται από διμερείς συμφωνίες που ε, χρονολογούνται το 1989. Οι βραζιλιάνικες αρχές χρησιμοποίησαν την διακριτική ευχαίρεια που προσφέρει ο νόμος για να απορρίψουν την αίτηση έκδοσης του Τσέζαρη Μπατίστη. Τονίζω εδώ με τρόπο σαφή ότι στην περίπτωση εκδόσεων δεν έχω αμφιβολία ότι η Ιταλική δικαιοσύνη θα σεβαστεί απολύτως τις υψηλές προδιαγραφές που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε περίπτωση εκδόσεως. Ευχαριστώ για το θέμα της εκδόσεως του Τσέζαρε Μπατίστη η συζήτηση έληξε. Έχω έξι προτάσεις ψηφισμάτων που θα ψηφιστούν μετά την ολοκλήρωση